σε μια ανακοίνωση από το Συμβούλιο έχω λάβει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση για την έγκριση του κανονισμού σε ό,τι αφορά την αλία στο πλαίσιο της συμφωνίας ε, GFCM, Γενικού Συμβουλίου Αλίας για ε, Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο θα δημοσιευθεί το σχετικό σημείο στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης ε, και από αύριο 11 Σεπτεμβρίου ξεκινά ε, η προθεσμία τριών μηνών που έχει στη διάθεση του Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη δική